Okay, colleagues, good... Λοιπόν, συνάδελφοι, καλησπέρα σα. Όπως ξέρετε, σκοπός συνέδρια είναι να συγκρατηθεί σε σώμα το Προεδρείο της Επιτροπής, υπό Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Θα εκλέξουμε πρώτα τον Πρόεδρο και κατόπιν τους Αντιπρόεδρους. Έχω και μια σειρά αναπληρωτών για τα τακτικά μέλη που απουσιάζουν. Από τα ΕΛΠ, ο κύριος Μικολάτσικ, θα αντικατασταθεί από τον κύριο Πέτερλε. Και, ο κύριος Αντάκτουσον επίσης απουσιάζει και θα αντικατασταθεί, αλλά δεν ξέρω από ποιον, από ποιον συνάδελφό του, από το ΕΛΚ θα αντικατασταθεί. Τώρα, ο κύριος Κάρσκι από τους συντηρητικούς μεταρρυθμιστές θα αντικατασταθεί από τον κύριο Τάνοκ. Ο κύριος Στάνοκ είναι παρόν. Από την άλλη ο κύριος Γκέρενς θα αντικατασταθεί από την κυρία Σάκη. Δεν ξέρω, μπορεί να κοιτάω σε λάθος κατεύθυνση, αλλά πού κάθεται η Άλντε, πού κάθονται οι φιλελεύθεροι. Α, γιατί δεν βλέπω την κυρία Σάκη που καθεται η αλντε που κάθεται οι φιλελευθεροι γιατι δεν βλεπω την κυρια σακη που αναπληρωνει τον συνάδελφό της από τους φιλελεύθερους. Από την ΚΟΕ, παρακαλώ ενημερώστε μας μου είπατε ότι ο κύριο Ιγκλέσια του Ριών ε, θα αντικατασταθεί από κάποιο για τη συνεδρίαση αυτή, αλλά δεν ξέρουμε από ποιον. Η κυρία Μαρίνα Αμπιόλς κανονικά έπρεπε να τον αναπληρώσει. Μάλιστα. Και για τους πράσινους, ο κύριος Μπίχνερ αντικαθίσταται από την κυρία Σαρχεντίνη. Άλλες αλλαγές υπάρχουν για το ΕΛΚ τουλάχιστον ή για κάποιο άλλο κόμμα. Όχι κανείς. Αυτές είναι οι αντικαταστάσεις. Μπορούμε να ψηφίσουμε τώρα. Να ελέγξουμε την απαρτία μας πρώτα. Οκτώ μέλη απαιτούνται για τη συγκέντρωση της απαρτίας. Βλέπω ότι έχουμε απαρτία. Υποψηφιότητες τώρα. Για τη θέση του Προέδρου. Κύριε Χάουιτ από τους Σοσιαλιστές, παρακαλώ, ποιος είναι υποψηφιό σας. Ευχαριστώ. Παρόλο που είναι επίσημη και τυπική αυτή η δήλωση. Με ιδιαίτερη χαρά θα ήθελα να προτείνω την κυρία Ελένα Βαλανσιάνο. Είμαστε και πάλι φίλοι και συνάδελφοι εκτός από την υποψήφια και αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά Ελένα για την υποψηφιότητά σου και σε θυμόμαστε παλιά σου συντονίστρια στην Επιτροπή μεταξύ 99 και στην επόμενη κοινοβουλευτική θητεία. Στη συνέχεια επέστρεψες ε, στο Εθνικό σου Κοινοβούλιο ήταν εκπρόσωπο των Σοσιαλιστών στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Και τώρα επανήλθε, επανέκαμψε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μα μεταδώσει το πάθο τη την προσήλωσή τη, την ακαιρεότητά τη για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ισότητε. Είναι αναφίβολη αυτή η προσήλωσή της και πιστεύω ότι θα ασκήσει την Προεδρία με πολύ δίκαιο τρόπο και χωρίς να αποκλεί κανέναν. Και με ιδιαίτερη χαρά προτείνω την υποψηφιότητά της για την Προεδρία της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κυρία Βαλενσιάνο, αποδέχεστε την υποψηφιότητα. Μάλιστα, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχουν άλλοι υποψήφοι για τη θέση του Πρόεδρου. Όχι, οπότε... Έχω και άλλες ερωτήσεις κυρία Βαλενσιάνο. Είστε τακτικό μέλος της Επιτροπής και φαντάζομαι ότι έχετε, έχετε υποβάλει τη δήλωση ε, οικονομικών συμφερόντων το πόθεν έσχεση. Έτσι. Μάλιστα. Οπότε μπορούμε να ψηφίσουμε διαβόηση. Και ελάτε κυρία Βαλενσιάνο να αναλάβετε την Προεδρία. Pues muchísimas gracias. Σας ευχαριστώ θερμά. Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που θέσατε την Προεδρία αυτής της Επιτροπής, της Υποεπιτροπής, με ιδιαίτερη τιμή και μεγάλη ευθύνη θα προεδρεύσω και μάλιστα αυτή την τιμή τη δέχομαι με ταπεινοφροσύνη και με την επιθυμία να συνεργαστούμε στενά όλοι προκειμένου να υλοποιήσουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για αυτή την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που έχει αυτόν τον τίτλο και τη συγκεκριμένη θέση στο οργανόγραμμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι υποεπιτροπή, αλλά για όλους εμάς, για όλα τα μέλη της, η Επιτροπή μας ε, δημιουργεί τεράστιες υποχρεώσεις και καθήκοντα. Γιατί τα ανθρώπινα δικαιώματα, η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να εξακολουθήσουν να βρίσκονται στο, στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής, εντός και εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μεριμνήσει και να δώσει το καλό παράδειγμα, να δίνει περισσότερο το καλό παράδειγμα παρά να κάνει κηρύγματα και να δίνει μαθήματα. Θα πρέπει αυτό όμως να τα επιδιώξουμε από κοινού με τη συνεργασία μας και με το έργο μας στην Επιτροπή αυτή. Στενή, άμεση και ειλικρινή συνεργασία μεταξύ όλων των πολιτικών ομάδων και φυσικά σε συντονισμό με τις υπόλοιπες ε, κοινοβουλευτικές επιτροπές με τις οποίες θα πρέπει να συνεργαστούμε για να προωθήσουμε το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων ε, όλων των συνανθρώπων μας ε, που διώκονται στις διάφορες περιοχές του κόσμου. Ε, σας διαβεβαιώ ότι το γραφείο μου θα είναι ανοιχτό και το τηλέφωνο μου ανοιχτή γραμμή για όλους έχουν κάποια ανάγκη, κάποιο σχόλιο ή κάποια ιδέα να προτείνουν είστε όλοι ευπρόσδεκτοι και θα ήθελα εκ των προτέρων να ευχαριστήσω τα Γραμματεία για τη συνεργασία και να την ευχαριστήσω για το, για το έργο που έκανε για την προετοιμασία αυτής της Επιτροπής. Περνάμε τώρα στην ε, εκλογή των αντιπροέδρων της ε, Επιτροπής μας. Αρχής γενομένης από τις πρώτες ε, υποψηφιότητες και θα ήθελα να ρωτήσω τις πολιτικές ομάδες ποιες υποψηφιότητες έχουν να καταθέσουν. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχήν να σας ε, συγχαρώ για την εκλογή σας και εκ μέρους ε, του Λαϊκού Κόμματος να σας συγχαρώ για αυτή τη σημαντική θέση. Σε αυτή τη τόσο σημαντική επιτροπή που είναι επιφορτισμένη με την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μετά την ε, συνθήκη της Λισαβόνας η Επιτροπή μας απέκτησε μεγαλύτερη σημασία. Θα ήθελα εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος να προτείνω για τη θέση του πρώτου Αντιπροέδρου τον συνάδελφό μας Κρίστια Πρέντα που ήταν και στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία Ευρωβουλευτής και εργάστηκε για τα θέματα αυτά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μάλιστα ήταν ε, εκπρόσωπο τη επικεφαλή τη Ρουμανικής Αντιπροσωπείας στο ΕΛΚ. Πολύ καλή υποψηφιότητα και η εμπειρία του θα εμπλουτίσει το έργο της Επιτροπής και θα βοηθήσουν την Επιτροπή στις εργασίε της. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, απευθύνομαι στον κύριο Πρέντα. Είστε πρόθυμος να δεχτείτε την υποψηφιότητα και να γίνετε μέλος του Προεδρείου. Είστε τακτικό μέλος φαντάζομαι της ε, Υποεπιτροπής και έχετε εκπληρώσει τις τυπικές προϋποθέσεις, έχετε καταθέσει το ποθενέσχες, πολύ ωραία. Άλλες υποψηφιότητες υπάρχουν για την πρώτη αντιπροεδρία της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όχι, οπότε αν γίνεται Ας εκλέξουμε διαβοής τον κύριο Πρέντα. Ελάτε παρακαλώ στο Προεδρείο. Έχουμε εκλέξει τον, πρώτο μας αντιπρόεδρο. Ποιες είναι οι υπόλοιπες υποψηφιότητες για δεύτερο αντιπρόεδρο ή αντιπρόεδρο γυναίκα, άντρα γυναίκα. Παρακαλώ. Θα ήθελα και εκ μέρου των φιλελευθέρων να σας συγχαρώ για την εκλογή σας και να πω ότι θα ήθελα να προτείνω την Μάουρα Μπαραντιαράν, που ήταν εκπρόσωπος του κόμματος για θέματα εξωτερικών υποθέσεων για πολλά χρόνια και είναι κατάλληλος υποψήφιος για τη θέση αυτή. Ελπίζω και προσβλέπω στην υποστήριξή σας για να υπερψηφίσουμε τον συνάδελφο στην ψηφοφορία για τη θέση του δεύτερου αντιπροέδρου. Κύριε Μάουρα, Είστε τακτικό μέλος της Επιτροπής, της Υποεπιτροπής. Μάλιστα, κυρία Πρόεδρε. Έχετε καταθέσει τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων. Μάλιστα, κυρία Πρόεδρε. Και θέλετε να γίνετε μέλος του Προεδρείου. Ε, με μεγάλη χαρά. Μάλιστα. Οπότε μπορούμε να εκλέξουμε τον κύριο Μάωρα που είναι παλιός ε, γνώριμος. Cumplimentada la elección del segundo vicepresidente. Τώρα για τον τρίτο αντιπρόεδρο. Ποιο είναι υποψήφιο, Κυρία Πρόεδρε, εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο θα ήθελα να προτείνω για τη θέση του τρίτου αντιπρόεδρου της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τον κύριο Λάσλο Τόκες. είναι Ούγγρος Ευρωβουλευτής και μάλιστα στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία ήταν μέλος της, Επιτροπής, της Υποεπιτροπής και μάλιστα συντονιστής ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Και μάλιστα ο κύριος ε, Λασλοτόκες έδωσε μεγάλη μάχη για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον εκδημοκρατισμό στη Ρουμανία. Και Ε, συνέβαλε στις ε, μεγάλες ε, πολιτικές αλλαγές που έγιναν στη Ρουμανία, λέει ο κύριος Ξύπ. Οπότε, με ιδιαίτερη χαρά θα ήθελα να προτείνω την υποψηφιότητά του. Ευχαριστούμε κύριε Τόκες. Είστε τακτικό μέλος της Επιτροπής. Έχετε εκπληρώσει τις τυπικές προϋποθέσεις ε, για τη συμμετοχή στο Προεδρείο και επιθυμείτε τη θέση αυτή. Οπότε αν δεν υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες, ε, να ψηφίσουμε διαβοής και τον τρίτο μας αντιπρόεδρο. Bueno, cumplimentada la elección de nuestro vicepresidente Μάλιστα, συγχαρητήρια και στον τρίτο μας αντιπρόεδρο. Και περιμένω την υποψηφιότητα του τέταρτου αντιπρόεδρου. Ποια ομάδα θα τον προτείνει. Thank you, Chair. It's... Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Με ιδιαίτερη χαρά θα ήθελα να προτείνω την κυρία Μπάρμπαρα Λοχμπίλερ για τη θέση της τέταρτης αντιπροέδρου. Είναι περί οι είναι γνωστή και η Βάρβαρα και η εμπειρία της στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με ιδιαίτερη χαρά θα τη δούμε να κάθεται στο Προεδρείο δίπλα σας. Ωραία. Βάρβαρα, εσύ έχεις τηρήσει τις τυπικές προϋποθέσεις, είσαι τακτικό μέλος της Υποεπιτροπής, θέλεις να λάβεις μέρος στο Προεδρείο. Ωραία. Αν δεν υπάρχουν άλλε υποψηφιότητε, προτείνω διαβοής να ψηφίσουμε και την τέταρτη πρόεδρο μας, την κυρία Λόχμπιλερ. Bueno, eh, ahora... Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, δύο μόνο ανακοινώσεις έχω να σας κάνω. Ανακοίνωση πρώτη. Το χρονοδιάγραμμα. Θα φροντίσουμε να συνεδριάσει το Προεδρείο μαζί με τους συντονιστές στο Στρασβούργο την άλλη εβδομάδα και προτείνω σε εκείνη τη συνεδρίαση να ορίσουμε και το χρονοδιάγραμμα το οριστικό, δηλαδή να καταλήξουμε. Νομίζω ότι θα πρέπει αυτό να συνάδει με τα θέματα που θέλουμε να συζητήσουμε. Πιο σημαντικό είναι να πούμε γιατί θέλουμε να μιλήσουμε και μετά να δούμε πότε θα συζητήσουμε γι' αυτό. Θα βρούμε, ε, ψάχνουμε ένα ε, χρονικό διάστημα για να συνεδριάσουμε στο Στρασβούργο λοιπόν και θα αποφασίσουν οι συντονιστές και το Προεδρείο για να δούμε ποια θέματα θα μας απασχολήσουν και μετά Οπότε, σε ό,τι αφορά το γλωσσικό καθεστώς, και πάλι θα το δουν αυτό οι συντονιστές με το Προεδρείο, γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι καθόλου οριστικό. Αυτές είναι λοιπόν οι δύο ανακοινώσεις που έχω να σας κάνω, οπότε όλοι θα ειδοποιηθείτε για ε, το χρονοδιάγραμμα τις ερχόμενες εβδομάδες. Δεν ξέρω αν έχετε τίποτα να πείτε, να ρωτήσετε. Ε, μια τοποθέτηση, ο Ρίτσαρτ Χάουιτ. Ναι. Συγγνώμη που σε διακόπτω και πάλι επειδή είμαι από άλλη πολιτική ομάδα, θέλω να το πω, εγώ ήμουν και στο παρελθόν βουλευτής, θέλω να αποτίσω ένα φόρο τιμή στην Μπάρμπαρα Μπίλερ ε, που ήταν σπουδαία πρόεδρος και ξέρω ότι θα είναι ε, εξίσου άξια και σπουδαία παραστάτη στο πλευρό σου το επόμενο διάστημα και όλους τους αντιπροέδρους θέλω να συγχαρώ που πιστεύω στο όνομά μας θα κάνουν μια καταπληκτική δουλειά. Uh, Κύριε Στάνοκ, θέλω και εγώ να προσθέσω τη φωνή μου σε εκείνη του Ρίτσαρτ Χάου. Είμαι ίσως από τους παλαιότερους εδώ στην Επιτροπή. Ο Ρίτσαρτ και εγώ διατελέσαμε πριν από μια οκταετία, αν δεν απατώ, με αντιπρόεδροι εδώ. Και τώρα είμαστε στα ορεινά βέβαια έδρανα, αλλά θα ήθελα να συγχαρώ όλους ε, και την κυρία Λοχμπίλερ και τους ε, άλλους αντιπροέδρους, εξ ονόματος μιας ομάδας που δεν έχει την Πρόεδρο, αλλά μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το τι συζητάει αυτή η Επιτροπή. Παραμένω αναπληρωτής, είμαι μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών, ακόμα και αν είμαι στα πολύ διαφορετικές πολιτικές παρατάξεις και οικογένειες, πρέπει να εξάρω το ρόλο της κυρίας Λόχ Μπίλερ. Συμφωνώ κι εγώ και φυσικά να ευχηθώ καλή επιτυχία στον εκλεγέν μας Προεδρείο και Νομίζω ότι είναι πολύ καλή συνήθεια αυτή να ξεκινάμε με συγχαρητήρια. Δημιουργεί ένα πολύ καλό κλίμα με τέτοια κατάσταση για το μέλλον της συνεργασίας μας. Επίσης θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συνεργασία που είχαμε στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα στην κυρία Μπάρβα Λοχμπίλερ. Ήμουν πρώτο αντιπρόεδρο στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία και πραγματικά θα ήθελα να ευχαριστήσω ολόθερμα την ε, κυρία Λόχμιλερ, για την Προεδρία που άσκησε στην προηγούμενη θητεία. Καλώς, νομίζω ότι ε, καλά τα πήγαμε. Σας ευχαριστώ όλους για τη συνεργασία σας που είμαι βέβαια ότι θα διατηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας. Σας ευχαριστώ πολύ και θα τα πούμε λίγαν συντόμως.